ταυτόχρονα ζητήσει με τη διαδικασία του catch Να λάβετε υπόψη σας ότι θα το συνυπολογίσω αυτό ως κριτήριο αν κάποιος κάνει χρήση της μπλε κάρτας ενδεχομένως να μην προτιμηθεί για τη διαδικασία του catch Το λόγο έχει ο κύριος Βάντε Ντρίσκε για ένα λεπτό. συνάδελφοι, τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ουγγαρίας και της Πολωνίας δεν έχουν να κάνουν με τα θέματα. Γιατί η μια χώρα όπως το Βέλγιο ε, με τα επιδοτούμενα μέσα ενημέρωση θα έπρεπε να έχει δεχτεί κυρώσει εδώ και καιρό. Το θέμα είναι ότι θέλουν να διατηρήσουν την ταυτότητά τους και την επικυριαρχία τους. Ποιος μπορεί να τους κατηγορήσει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή μπορεί να δίνει λύσεις και δεν δίνει λύσει, μάλλον ούτε για την ε, κρίση του ευρώ, ούτε για την κρίση τη μετανάστευση. Η ελίτα δεν δίνει λύσεις. Ε, επιβάλλει από πάνω προς τα κάτω νόμους. Καταστρέφεται λοιπόν την Ευρώπη με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση των δικτατόρων και των γραφειοκρατών. Με το Brexit έχουμε την πρώτη χώρα η οποία θα αποχωρήσει. Πόσες χώρες πρέπει να βγουν για να καταλάβετε ότι πρέπει να... επιτέλους να ακούσετε τον κόσμο. Ένα λεπτό κύριος Λούντγκρεν. Ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζω ότι οι σοσιαλιστές και δημοκράτες έχουν διαφορετική άποψη για την Ουγγαρία και την Πολωνία. Η Ουγγαρία είναι κυρίαρχο δημοκρατικό κράτος και ε, πρέπει να έχει την ε, δυνατότητα ε, αυτοδιάθεσης εντός των δημοκρατικών διαδικασιών. Υπάρχουν πολλές χώρες που τις πιάνει η ιστερία και αρχίζουν και φωνάζουν ότι συμβαίνουν σκάνδαλα τρομερά και φοβερά. Ωστόσο, ε, είναι γεγονός ότι η κάθε χώρα έχει δικαίωμα στην αυτοκυριαρχία και στο να αποφασίζει μόνη της ε, τον τρόπο με τον οποίο θέλει να κυβερνιέται. Όταν ε, θέλουμε, ας πούμε, να μειώσουμε τα εθνικά σύμβολα, υπάρχουν χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως που δεν μπορούν να το δεχτούν αυτό. Εδώ όλοι επιθυμούν ε, ε, να εκπροσωπούνται ε, σαν να ήταν στα εθνικά κοινοβούλια. Θα ήθελα να ε, αποτίσω φόρο τιμή ε, για τον Ρότζερ Χάρτμαν, τον Άγγλο φιλόσοφο και φίλο μου, ο οποίος ε, πέθανε αυτή την εβδομάδα. Υπάρχουν χώρες όπως η Ουγγαρία και η Πολωνία που προσπαθούν να ανακτήσουν την κυριαρχία τους μετά από την επικυριαρχία της Σοβιετικής Ένωσης. Ε, η Πολωνία και η Ουγγαρία έχουν την δυνατότητα και την υποχρέωση απέναντι στους πολίτες τους να παίρνουν τέτοιες ε, αποφάσεις και δεν είναι δυνατόν να υποκύπτουμε ε, σε ολοκληρωτισμούς και τέτοιου είδους συμπεριφορές. Ούτως ή άλλως ε, είμαστε διαφορετικοί, έχουμε διαφορετικά εκλογικά συστήματα, ε, θα πρέπει να ζήσουμε με αυτά. Εσείς ε, λέτε ότι από τη μία μεριά ότι θέλετε την διαφορετικότητα, από την άλλη μεριά όμως απαγορεύετε στους ανθρώπους να σκέφτονται διαφορετικά και να σκέφτονται με άλλο πολιτικό τρόπο. Δεν, και, και ξεκινάτε διαδικασίες επί παραβάση για όσους δεν σκύβουν το κεφάλι. Έχει ο κύριος Ρανζέλ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έκαναν το καθήκον τους. Μπράβο σας. Θα ήθελα να επιθυμίσω το βασικό, ότι ε, η Ευρώπη είναι μια λέσχη δημοκρατίας ε, που σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη διάκριση των εξουσιών και το κράτος δικαίου. Και γι' αυτό κάθε φορά που υπάρχει ε, μία παραβίαση αρχών του κράτους δικαίου και έλλειψη σεβασμού στους πυλώνες της δημοκρατίας μας, θα πρέπει να ε, εφαρμόζεται ο μηχανισμός για να εξακριβώνεται αν τα κράτη-μέλη ε, εφαρμόζουν αυτές τις αρχές. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα με την Ουγγαρία, υπάρχουν προβλήματα με την Πολωνία, ακόμη και με τη Μάλτη υπάρχουν προβλήματα. Είναι αλήθεια όμως ότι το άρθρο 7 δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε και γι' αυτό είναι κέρια σημασία στη συζήτηση αυτή να προασπίσουμε και να προτείνουμε ένα μηχανισμό που θα μπορεί να ελέγχει και να εξακριβώνει, να επαληθεύει την εφαρμογή των κανόνων του κράτους δικαίου σε όλα τα κράτη-μέλη, χωρίς διακρίσεις και χωρίς ε, να δίνεται εντύπωση ότι υπάρχει δίωξη συγκεκριμένου κράτους. Ελπίζω οι κυβερνήσει τη Ουγγαρία και τη Πολωνία να κάνουν κάποια θετικά βήματα πρόοδου και να δώσουν κάποια ε, σημάδια σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του άρθρου 7. Ευχαριστώ. Αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, αν ήσταν αρκετά φίλοι για να πιστεύετε ότι η έκθεση Αρχεντίνη θα σταματήσει τον Βίκτορ Όρμπαν, τι να πω. Κάνετε λάθος. απατάστε. Φαίνεται ότι συνεχίζει ακάθεκτος ο Όρμπαν επιτίθεται στα δικαστήρια, επιτίθεται στην πολυφωνία των ΜΜΕ. Έχει ε, κλείσει τα ανεξάρτητα θέατρα. Μόνο τους πιστούς και αφοσιωμένους του προστατεύει και μάλιστα θέλει να συγκεντρώσει την κατανομή των κοινοτικών κονδυλίων αφαιρώντας τη σχετική εξουσία από την τοπική αυτοδιοίκηση. Επίσης έχουμε έναν ε, συμπολίτη μας που ήταν ε, απλός βιοπαλαιστής και τώρα έχει γίνει πολυεκατομμυριούχος. Ο κύριος Όρμπαν καταστρατηγεί τις ευρωπαϊκές αξίες και χρησιμοποιεί τα κοινοτικά κονδύλια για να χρηματοδοτεί τις εκστρατείες του εις βάρος των ευρωπαϊκών αξιών. Αν δεν σταματήσουμε εμεί τον Όρμπαν, μόνος του αποκλείεται να υπαναχωρήσει. Και αν απλώς ε, εκφράζουμε την ανησυχία μας, τη θλίψη μας ε, ε, για τα τεκτενόμενα στην Ουγγαρία και απλώς συντάσσουμε μακροσκελείς εκθέσεις, δεν θα κάνουμε τίποτα. Ο Όρμπαν δεν καταλαβαίνει τα λόγια. Το μόνο που καταλαβαίνει είναι η βία, η αποφασιστικότητα, η πυγμή. Θα πρέπει να του πούμε σταμάτα να ξοδεύεις τα κοινωτικά κονδύλια σαν να είναι ιδιωτικά σου χρήματα. Μόνο με τιμωρία καταλαβαίνει ο Όρμπαν. Μόνο έτσι θα προστατεύσουμε τους Ούγκρους και θα προσπίσουμε τα συμφέροντα του Ουγγρικού λαού. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι πολίτες στην Ουγγαρία υπόκεινται σε διακρίσεις. Τα παιδιά από τις οικογένειες Ρωμά διώκονται και δεν μπορούν να διαβάσουν αυτά τα παιδιά αφού τελειώσουν τη σχολική του εκπαίδευση. Ουσιαστικά δεν έχουν πραγματική εκπαίδευση. Την προηγούμενη εβδομάδα ένα δικαστήριο έδωσε αποζημίωση στις οικογένειες αυτές για την κοινωνική απομόνωση και δικαίω γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτή η θεσμική, ο θεσμικό ρατσισμό στην Ουγγαρία. Πώ αντιδρά λοιπόν ο κύριο Ορμπάν, αντί να προστατεύσει τα παιδιά αυτά, φροντίζει να απομονωθούν πιο πολύ και εκ νέου πρόχνει ε, και προωθεί τον αντιτσιγκανισμό, τον ρατσισμό. Κύριε Ορμπάν, σταματήστε να διαδεδετε κατά των ε, τσιγκάνων των μειονοτήτων και εσείς ε, αξιότιμοι κύριοι του Τσεντεού, ε, επιτέλους ε, κλείσετε, ε, διώξτε τον Ορμπάν από την οικογένειά σας και επιτρέψτε στο άρθρο 7 να τιμωρήσει σωστά τον κύριο Ορμπάν. Έχετε μπλε κάρτα, κυρία Φράντσα, από την κυρία Γιάροκα και, έχουν και άλλα, υπάρχουν και άλλα αιτήματα για ερωτήσεις στην μπλε κάρτα. Τη δέχεστε? Έχετε το λόγο για 30 δεύτερα, κυρία Γιάροκα. Σας ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε, που δεχτήκατε αυτή την μπλε κάρτα και ξέρετε ότι συνεργαζόμαστε πολύ στενά για το θέμα των Ρωμά. Γι' αυτό, λοιπόν, θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω, Ρωμαίο, πείτε μας άλλη μια χώρα που έχει κάνει πιο πολλά για τους Ευρωπαίους Ρωμά από ότι η Ουγγαρία. Πείτε μου μία μόνο χώρα που να έχει κάνει πιο πολλά για τους Ευρωπαίους Ρωμά από ότι Ουγγαρία. Σας παρακαλώ. Liebe Livia, Αγαπητή Λίβια, αυτή η ερώτηση δεν είναι καν σωστή. Θα ήθελα... Θα ήθελα... Αυτά τα οποία διατείνεστε να ήταν αληθινά, μακάρι. Αλλά έχουμε αποτεκτικά στοιχεία, γεγονότα τα οποία πιστοποιούν ότι πριν από κάποιε ημέρε αυτή η δικαστική απόφαση πιστοποιεί. Αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί, είναι η αλήθεια. Ας μιλήσουμε λοιπόν με, για συγκεκριμένα γεγονότα, για το πώς μπορούμε αυτή την κατάσταση να την αλλάξουμε για τους ανθρώπους αυτούς. Αυτό δεν κάνουμε και οι δύο. Προσπαθούμε αυτό να πετύχουμε, αλλά δεν μπορούμε να το πετύχουμε βάσει ψεμάτων. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα αποδεκτικά στοιχεία, τα δεκμήρια και να προσπαθήσουμε όλα αυτά να τα αλλάξουμε. Αυτή είναι η προσέγγιση που ακολουθούμε. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Τσαμπάτσκι για ένα λεπτό. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η διαδικασία ε, ε, ενάντια στην Ουγγαρία και την ε, Πολωνία δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς γιατί έχει ξεκινήσει. Γιατί οι Πολωνοί και οι Ουγγροί ε, ε, εκλογής με ελεύθερο και δημοκρατικό τρόπο ε, επέλεξαν την κυβέρνησή τους. Ε, αυτοί που προτιμούν ε, τα κόκκινα κομμουνιστικά ε, σύμβολα από τα εθνικά σύμβολα δεν τους αρέσουν αυτά που γίνονται ή λέγονται ή στην Ουγγαρία για τα σύνορα ή για τους μετανάστες. Δεν σας αρέσει αυτός ο τρόπος, αλλά στην ουσία εσείς φέρεστε σαν Πολσεβίκοι, σαν δικτάτορες και αρνείς τους ε, ε, Πολωνούς και Ούγγρους ε, πολίτες να αποφασίζουν ελεύθερα για την μοίρα τους. <clears throat> Πολλές αυτοκρατορίες προσπάθησαν να σταματήσουν τον κόσμο από το να αποζητά την εθνική του ταυτότητα, δεν τα κατάφεραν. Μπλε κάρτα από την κυρία Μπάρλεϊ, τη δέχεστε. Η κυρία Μπάρλεϊ έχει το λόγο. Do you, Συμφωνείτε ίσως μαζί μου ότι οι δικτάτορες προσπαθούν να ελέγχουν πάντα όλες τις εξουσίες και αυτό το κάνετε κι εσείς ε, και ε, συμφωνείτε ότι αυτό ακριβώς συμβαίνει τούτη τη στιγμή στην Ουγγαρία. Κύριε Τσαμπάσκι, 30 δεύτερα. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφε, αυτό που είπατε δεν συμβαίνει στην Ουγγαρία. Οι πολίτες στην Ουγγαρία και την Πολωνία εξέλεξαν την κυβέρνησή τους. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι όταν εσείς δεν συμφωνείτε μαζί μας, δεν μας δίνετε τη δυνατότητα, δεν μας αφήνετε να μιλάμε. Αυτό ε, αποτελεί ε, απομείωση της ελευθερίας μας. Αυτό είναι ο βολσεβισμός ακριβώς. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Μπελαμή. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, συμφωνούμε όλοι εδώ ότι θα πρέπει να υπερασπιστούμε το κράτος δικαίου γιατί αυτό είναι ουσιώδες. Αλλά τι συμβαίνει, τι συμβαίνει στην Ουγγαρία, είναι ελεύθερες οι εκλογές, ναι. Υπάρχουν, υπάρχει πολιτικός πλουραλισμός, ναι. Ε, το, τα μέσα ενημέρωσης έχουν την δυνατότητα να ασκήσουν κριτική. Από ό,τι ξέρω δεν έχει δολοφονηθεί κανείς ε, δημοσιογράφος. Δεν είδα όμως την ίδια ζέση πριν από λίγο καιρό όταν συζητούσαμε για το ίδιο θέμα. Λοιπόν, μπορούμε ε, να συνεχίσουμε, αν θέλετε, μπορούμε να συνεχίσουμε ε, να προσβάλλουμε την επιλογή των ε, πολιτών των χωρών αυτών. δεν έχουμε την δυνατότητα όμως οποιαδήποτε πολιτική μας αντίθεση να την μεταφέρουμε ε, σε μια συζήτηση που θα αφορά το κράτος δικαίου. Δεν είναι δυνατόν να το κάνουμε αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Μπελαμή, έχετε ε, μία μπλε κάρτα από ένα μέλος της δικής σας πολιτικής ομάδας, την κυρία Τούν, τη δέχεστε? Κυρία Τούν, παρακαλώ. 30 δεύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε, από τη δική μου πολιτική ομάδα. Θα ήθελα να ρωτήσω οι εκλογές είναι πραγματικά ελεύθερες όταν τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι ελεύθερα. Δεύτερη ερώτηση. Πρέπει πραγματικά να δολοφονηθεί ένας δημοσιογράφος για να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει ελευθερία του τύπου. Τρίτον, η κυβέρνηση ακόμα και αν έχει εκλεγεί από την πλειοψηφία των εκλογέων έχει δικαίωμα να δρά κατά της δημοκρατίας, κατά της δικαστικής εξουσίας, κατά του κράτους δικαίου. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. An Ενδιαφέρουσες αυτές οι ερωτήσεις. Έχετε 30 δευτερόλεπτα, κύριε συνάδελφοι από την ίδια πολιτική ομάδα. Τρει απαντήσει, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, υπάρχουν ε, μέσα ενημέρωση ε, που αντιτίθενται και επικρίνουν την κυβέρνηση. Δεύτερον, ναι, όταν ένας δημοσιογράφος δολοφονείται, ναι, είναι μεγάλο πρόβλημα και δεν υπάρχει σε αυτή την περίπτωση ενεργοποίηση του άρθρου 7. Ε, ε, κοιτάξτε, εσείς ε, μιλήσατε προηγουμένως άσχημα για μένα. με βρίσατε στην ουσία. Είπατε ότι είναι ντροπή που παίρνω το λόγο. Ε, απ' την άλλη πλευρά δεν είναι δυνατόν οι διαδικασίες οι οποίες προδίνουν τον κόσμο να μας βρίσκουν σύμφωνους. Ε, κύριε Μπελαμή, λέει ο Πρόεδρος, ε, σύμφωνα με τον κανονισμό ε, είχατε 30 δευτερόλεπτα για να απαντήσετε στην ερώτηση της κυρίας Τούνη και όχι σε άλλες ερωτήσεις άλλων συναδέλφων. Παρακαλώ πολύ να σέβεστε τον Πρόεδρο και να ακολουθείτε τους κανόνες. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Ζίπελ. Ευχαριστώ πολύ και πάλι η Ουγγαρία, οι διαμαρτυρίες της αντιπολίτευσης, ε, θέματα στο πολιτισμικό το προσκήνιο, ό,τι και να συμβαίνει δεν μας απασχολεί. Όπως και παλιά στην Ουγγαρία έχουμε ένα ακόμα και μία άποψη. Στο μέλλον η, Ευρω... η κυβέρνηση θέλει να αποφασίζει πόσα χρήματα θα παίρνουν οι δημικοί κοινότητες και πώς θα διορίζονται οι αξιωματούχοι. Το νέο πολιτισμικό λοιπόν συμβούλιο θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για τέτοια ζητήματα. Δεν μπορεί να είμαστε όμως αφελείς. Ο πολιτικός έλεγχος των ε, πολιτισμικών ε, θεσμικών οργάνων φτάνει στα όρια της λογοκρισίας και οι αποκλίνουσες απόψεις δεν πρέπει καν να ακούγονται, να μην υπάρχει πλατφόρμα για, αυτέ. για αυτές. Ε, και παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει καμία σαφή απάντηση από την Επιτροπή και από το Συμβούλιο. Η νέε εξελίξει, οι μη δημοκρατικές εξελίξεις στην Ουγγαρία δεν ε, γίνονται αποδεκτέ προφανώς από τον κόσμο. Είναι σκανδαλώδε. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρξουν σαφείς συνέπειες πλέον. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Σκοτ Κάτω. Thank you, President. Ευχαριστώ. Η αναπτυσσόμενη σύγκληση μεταξύ της Βρετανικής κυβέρνησης και του Βίκτορ Όρμπαν θα πρέπει να χτυπάει καμπανάκι για όλους τους δημοκράτες. Καταρχήν, ε, ζητήθηκε ειδική σχέση Ουγγαρίας-Βρετανίας και ο Όρμπαν επενεί τον ε, Τζόνσον ως το, το, το γενναιότερο από τους γενναιότερους πολιτικούς. Ε, αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνούμε όταν διαπραγματευόμαστε τι μελλοντικέ μα σχέσει με το Ηνωμένο Βασίλειο. Μήπω θα γίνει μια ψευτοδημοκρατία το Ηνωμένο Βασίλειο κατά το ουγγρικό πρότυπο. Από το 2010 η κυβέρνηση Όρμπαν επιτίθεται κατά τη ελευθερία ε, των ΜΜΕ, περιόρισε το, την πρόσβαση μη φίλων δημοσιογράφων, αφαίρεσε την άδεια από το BBC και γενικώ ε, ε, έχει ακροτηριάσει την ελευθερία των ΜΜΕ. Αυτή είναι μια κατάσταση χειρότερη από ποτέ. Επίσης, ο Όρμπαν είναι υπέρ του Brexit, γιατί αποτελεί μια κίνηση της αυταρχικής κυβέρνησης και μάλιστα οι Τόρις ε, έστρωσαν κόκκινο χαλί για τον Ούγκρο ε, Πρωθυπουργό και αυτό είναι κρίμα και ντροπή όχι μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κάποιο στοιχείο ένωση συνεργασία, ούτε έχει κάποιου στοιχείου κανόνε. Είμαστε μια κοινότητα αξιών και όποιοι είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σέβονται τι ευρωπαϊκέ αξίε, ε, δημοκρατία, ελευθερία, ε, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά είναι η βάση τη συνεργασία, μα. Χωρί αυτά τα στοιχεία λοιπόν δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να επιμείνουμε τόσο πολύ για να τηρούνται αυτέ οι αξίε σε όλα τα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ στο Κοινοβούλιο, πριν από 1,5 χρόνο, διαπιστώσαμε ότι αυτέ οι αξίε διακυβεύονται στην Ουγγαρία. Εμεί το υποστηρίξαμε τώρα και τα τελευταία 1,5 έτος δεν μειώθηκαν οι λόγοι ανησυχία. Γι' αυτό λοιπόν είναι καλό αυτό που κάνουμε σήμερα, το γεγονό ότι αύριο θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε το ψήφισμα. Αλλά θα πρέπει η πραγματική συζήτηση να γίνει στου κόλπου του Συμβουλίου. Δεν γίνεται αυτό γιατί οι χώρε δεν τολμούν να συζητήσουν αυτό επαρκώ θα πρέπει λοιπόν να το πούμε προς τους αρχηγούς κρατών κυβερνήσεων. Δείξτε ότι και για σας το κρατός δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία είναι πιο πολλά πράγματα πέρα από τις α, όμορφες κουβέντες και την προεκλογική εκστρατεία. Το λόγο έχει η κυρία Ιντσίρ. there is a Μία μπλε κάρτα έχετε. Εκτός μικροφώνου. Δέχεστε την μπλε κάρτα. Ε, συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφο, αλλά ε, έχω ένα δίλημα και θα ήθελα να με βοηθήσει. Απ' τη μια πλευρά μιλήσατε εκ μέρου τη πολιτική ομάδα και είπατε ότι θα πρέπει να προσπίσουμε τι ευρωπαϊκέ αξίε και θα πρέπει να το συζητήσουμε. Και απ' την άλλη έχουμε Ούγγρου ε, συναδέλφου που καταστρατηγούν αυτές τις αξίες και τις αμφισβητούν. Θα συμφωνήσετε επιτέλους μεταξύ σας για να δούμε σε ποια πλευρά βρίσκεστε. Well, it's not my job to solve your Δεν είναι δική μου δουλειά να λύσω τα δικά σας διλήμματα. Μπορείτε να το κάνετε μια χαρά και μόνο σας. Εμείς συζητάμε αυτά στην ομάδα μας, τα συζητάμε αυτά στην οικογένειά μας. Θα τα συζητήσουμε και στο μέλλον προφανώς. Αυτά έχω να πω εγώ. Εσεί φροντίσετε τη δική σα ομάδα και συγχαρητήρια και καλή τύχη με του Μαλτέζου συναδέλφου του και εμεί θα συζητήσουμε τα δικά μα με τη δική μα ομάδα. Προχωρούμε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Το λόγο έχει η κυρία Ιντσίρ για ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ. Ο Βίκτορ Όρμπαν ενισχύει τις επιθέσεις του κατά της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ουγγαρία. Μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατάφερε να βρει μια λύση. Και στο μεταξύ έχει επιδεινωθεί σημαντικά η κατάσταση στην Ουγγαρία. Και αν υπήρχε βραβείο ευρηματικότητα και δημιουργικότητα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ούγγροι του Όρμπαν και οι Πολωνοί του Πις θα το κέρδιζαν. Γιατί έχουν πολύ ευρηματικού τρόπου για να επιτεθούν ε, στι θεμελιώδει αξίε και του κανόνε Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει μείνει ανενεργό το άρθρο 7. Θα πρέπει να βρούμε ένα νέο μηχανισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να προασπίσουμε σωστά το κράτο δικαίου, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και να προτείνουμε και επιβολή κυρώσεων όταν κράτη-μέλη καταστρατηγούν τι στοιχειώδει ε, διατάξει Ευρωπαϊκή Ένωση όπω το άρθρο 2. Θα πρέπει να μην έχουν πρόσβαση και στη χρηματοδότηση οι χώρε αυτέ. Δεν μπορεί να δέχονται οι Ευρωπαίοι πολίτε τα κοινοτικά κονδύλια να χρησιμοποιούνται ε, απρεπώς για να ασκείται επίθεση στις αξίες μας. Σα Σας ευχαριστώ. Ο σεβασμός των κοινών μας αξιών και του κράτους δικαίου αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους στις κοινωνίες μας. Βέβαια, ο τρόπος που αποτελούν κοινωνικούς κανόνες και πώς γίνεται ο έλεγχός τους είναι θέμα προσυζήτηση. Καλή ανταλλαγή απόψεων, αλλά αυτό που κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να κραδένει το φόβητρο του άρθρου 7 κατά της Ουγγαρίας, ενώ δεν υπάρχουν διατάξεις που να το προβλέπουν. Δεν θα πρέπει να εσφετεριζόμαστε τα δικαιώματα του Συμβουλίου της Επιτροπής και να μην υποβάλλουμε προτάσεις που υπερβαίνουν τις συνθήκες. Το κείμενο μιλά για φόβο υπονόμευσης των αξιών και ε, της τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν όμως ήδη ξεκινήσει δύο διαδικασίες ει βάρος δύο χωρών τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ υποτίθεται ότι όλε οι υπόλοιπε χώρες είναι μια χαρά. Έχουμε διπλά μέτρα και σταθμά. Αυτά είναι που υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά θα πρέπει να καταπολεμήσουμε. Για ένα λεπτό. Thank you, President. Ευχαριστώ. Πριν από 1,5 περίπου χρόνο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να ενεργοποιήσουν τη διαδικασία του άρθρου 7 κατά τη Ουγγρική κυβέρνηση. Και το μόνο που είδαμε έκτοτε είναι 1,5 χρόνο ε, ενδιασμών, διστακτικότητα στο Συμβούλιο και ε, μεταφέρουν την καυτή πατάτα από τη μία προεδρία στην άλλη. Ενώ ο Όρμπαν δεν διστάζει καθόλου. Είναι αδίστακτος ε, και εξακολουθεί να υπονομεύει την ανεξαρτησία των δικαστών, να καταστρέφει τον πλουραλισμό των ΜΜΕ και να υποδαβλίζει ξενοφοβικέ τάσει. Και εμεί τον αφήνουμε ενόχλητο. Το Συμβούλιο εξακολουθεί να μπλοκάρει την πρόοδο του άρθρου 7. Ε, Παρατηρήνω την Κροατική Προεδρία να λάβει σοβαρά υπόψη το άρθρο 7 και να το καταστήσει προτεραιότητα. Και διαρωτώ με συνάδελφοι, η αντιπροσωπεία του Φίντε στην επόμενη Ολομέλεια μήπως θα πρέπει να καθίσει πιο δεξιά, γιατί εκεί ανήκουν, στην ακροδεξιά. Πολλοί Ούγγροι εξακολουθούν να πιστεύουν στη δημοκρατία, εξακολουθούν να πιστεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο δικό τους πλευρό στεκόμαστε. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Χιτβέγγι. Σας ευχαριστώ. Για να δούμε γιατί κατασκευάστηκε αυτή η διαδικασία εις βάρος της Ουγγαρίας και της Πολωνίας. Αυτό συνέβη γιατί επέμειναν οι αριστερές πολιτικές δυνάμεις ε, να τεθεί η ενεργοποίηση του άρθρου 7 ως προϋπόθεση για να συζητηθεί η δολοφονία της Μαλτέζας δημοσιογράφου. Έτσι έγινε η συζήτηση τον Ιανουάριο. Είναι α, ε, ανεδαφικές όλες οι κατηγορίες βάρος Ουγγαρίας. Και δικαστική ελευθερία υπάρχει και ελευθερία λόγου και έκφρασης υπάρχει και τα ΜΜΕ ε, έχουν μια πολυμορφία και γίνεται συζήτηση στην Ουγγαρία, ακόμη και με τις αριστερές δυνάμεις Ευρώπης. Θέλουμε να προστατεύσουμε την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και ταυτόχρονα την εθνική μας κυριαρχία. Η κατάχρηση του κράτους δικαίου γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να τιμωρηθεί πολιτικά η Ουγγαρία και η Πολωνία με αυτή τη διασκευασμένη διαδικασία. Μπλε κάρτα, δέχεστε. Ευχαριστώ πολύ. Τι σπάνια στιγμή πολιτικός του Φίντες να μπει στη συζήτηση. Δεν έχει γίνει αυτό από τότε που έχετε βγει στην κυβέρνηση. Μία απλή ερώτηση. Αν ε, σύμφωνα με το Φίντες και τον ε, Ορμπάν όλα πάνε καλά με το κράτος δικαίου, γιατί είστε τόσο έντονα κατά της δέσμευσης ε, των ευρωπαϊκών πόρων με το κράτο δικαίου. Δεν είναι αυτό παραδοχή τη υπετιότητά ε, σα. 30 δεύτερα έχετε για να απαντήσετε. Ναι, ευχαριστώ. Ναι, αυτό ακριβώς συζητάμε. Ότι οι δυνάμει τη αριστερά ε, καταχρώνται τη ε, ιδέας, της αξίας του κράτους δικαίου και το κάνουν πολιτικό εργαλείο. Εσείς είσαστε οι αυτοί που είστε αντίθετοι στις ανεκτικότητες και του αντίθετη με τι αξίε ε, του λαού. Θέλουμε λοιπόν να ισχύουν όλα με του ίδιου όρου για όλου. Δεν συμβαίνουν αυτά τώρα. Χρησιμοποιήσετε το κράτο δικαίου για πολιτικό κυνήγι μαγισσών. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από παραπάνω από 1,5 χρόνο πριν το Κοινοβούλιο ε, ψήφισε επίσημω ε, την ενεργοποίηση του άρθρου 7 παράγραφος 1. Ε, όμως οι κυβερνήσει τη Ουγγαρία και τη Πολωνία εξακολουθούν να παραβιάζουν το κράτο δικαίου. Ε, εν τω μεταξύ έχουν ξεκινήσει συζητήσει μεταξύ εμπειρογνωμόνων, επιτροπών κλπ. Αλλά τίποτα. Και ούτω ή άλλω ε, τα ευρωπαϊκά κονδύλια εξακολουθούν να πλουτίζουν στηρίζουν τους φίλους ε, και τους ε, κοντινούς ανθρώπους του κυρίου Ορμπάν. Ε, θα πρέπει να είμαστε σοβαροί τουλάχιστον μεταξύ μας. Θα πρέπει να χτυπήσουμε εκεί που πονάει η χώρα. Θα πρέπει στη Βαρσοβία, στη Βουδαπέστη, παντού πολιτική, ακαδημαϊκή κοινότητα, νέοι φοιτητέ, μη κυβερνητικέ οργανώσεις κινητοποιούνται. Θα πρέπει να ε, που με ότι εντωμεταξύ ο κύριος Ορμπάν όλα αυτά τα οποία συζητιούνται τα κάνει χαλάκι για να καθαρίζει τα πόδια του. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο Χάνσεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το κράτος δικαίου ε, σημαίνει ότι το δίκαιο είναι αυτό το οποίο υπερισχύει ε, σε μια ε, δημοκρατική χώρα που συμμερίζεται τις δημοκρατικές αξίες τις οποίες σέβεται το, η Ευρωπαϊκή Ένωση ο ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας ε, λέει ότι ε, υπάρχουν, έχουν ληφθεί αποφάσεις οι οποίες αντιτίθενται στο σεβασμό της ε, ιδιωτικής ζωής, στον, στο δικαίωμα του συνεστερίζεστε, καθώς επίσης και στην ελευθερία κίνησης. Στην ουσία δηλαδή έχουμε διαρκώς επισοδρομήσεις, ένα βήμα μπρο, τρία βήματα πίσω, αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Σε όλα τα κράτη-μέλη και άσχετα από το τι χρώμα έχει η πολιτική εξουσία, θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να υπεραμεινόμεθα των δημοκρατικών αρχών. Το λόγο έχει η κυρία Φόλατ για ένα λεπτό. Έχετε το λόγο, κύριε Φόλατ. Στην ουσία και στην αλήθεια είναι συγκλονιστικό ότι η έκθεση του 2018 εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ε, είχε καμία σωστή αντίδραση από πλευρά τη ε, Ουγγαρία, ούτε από το Συμβούλιο προκάλεσε κάποια σωστή αντίδραση. Η Ουγγρική κυβέρνηση συνεχίζει να παραβιάζει το κοινωτικό δίκαιο ανεκτά και είναι όλο και πιο πολύ δημοκρατία μόνο στα χαρτιά, καταπιέζοντα την ε, ελευθερία του τύπου χωρί ε, ανεξαρτησία για τους μεγάλους θεσμούς, τα πανεπιστήμια, για όλου αυτού του θεσμού. και το Συμβούλιο απλά παρακολουθεί την κατάσταση. Οι εξελίξει αυτέ ε, σημαίνει, σημαίνουν ότι πρέπει να αφήσουμε κατά μέρο το ευρωπαϊκό έργο. Θέλουμε λοιπόν να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι μόνο να κινητοποιήσει το άρθρο 7 και να συνεχίσει την κινητοποίηση, αλλά και να ολοκληρώσει την νομοθεσία για την δέσμευση των ευρωπαϊκών πόρων με τους όρους του κράτους δικαίου. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των εγγεγραμμένων ομιλητών. Προχωρούμε στη διαδικασία του Catch the Eye. Έχω δεχθεί πέντε αιτήματα. Ένας από τους συναδέλφους που ζήτησε το λόγο με τη διαδικασία του Catch the Eye έχει κάνει χρήση ήδη του δικαιώματος της μπλε κάρτας. Επομένως, κάνω τα υπόλοιπα τέσσερα αιτήματα αποδεκτά. Το λόγο έχει η κυρία Γκιόρη για ένα λεπτό. Az Unióban világosak a szabályok és az intézmények közötti munka. Ευχαριστώ πολύ. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα διάφορα θεσμικά όργανα έχουν ξεκάθαρους ε, ρόλους. Ε, όμως ε, υπάρχουν στο κείμενο της πρωτοβουλίας της αριστεράς δύο ε, ασάφειες και το Συμβούλιο στη θέση του και η νομική υπηρεσία του ΕΛΚ λέει ότι υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τον, το ευρωπαϊκό δίκαιο. Απ' την άλλη πλευρά όμως δεν μπορούν να σταθούν αυτές οι γενικές κατηγορίες ε, σε σχέση με το άρθρο 7. Ε, κυρία Επίτροπε, νομίζω ότι θα ήταν πραγματικά ιδιαίτερα λυπηρό να επιμείνει η Κομισιόν στη διαδικασία αυτή. Δεν είναι δυνατόν να μπερδεύονται τα πολιτικά και τα ε, νομικά δικαστικά ζητήματα και νομίζω ότι το κράτος δικαίου και ο έλεγχος της εφαρμογής του κράτους δικαίου θα πρέπει να γίνεται με ίδιο τρόπο από όλους. Ο κύριος... Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Λόπες Αγγελάρ. Πριν από 10 χρόνια ο Βίκτορ Ορμπάν ε, ξεκίνησε ε, ε, την διακυβέρνηση της Ουγγαρίας με μεγάλη πλειοψηφία αλλά όμως επανέρχεται διαρκώς ξανά και ξανά το θέμα της Ουγγαρίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ ως πρόεδρος της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ προείδρευσα της πρώτης αποστολής που ασχολήθηκε με τα δικαιώματα των ε, μειοψηφί των μειονοτήτων, την ελευθερία της ακαδημαϊκής κοινότητας ε, και των μέσων ενημέρωσης, καθώς επίσης ε, μελετήσαμε και κάποιες καταγγελίες για διασπάθηση και διαφθαρά όσον αφορά την χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το θέμα δεν είναι πάντα ε, ε, το, το θέμα δεν είναι πάντα ε, η κυβέρνηση που έχει εκλεγεί δημοκρατικά να έχει πάντα δίκιο. Το θέμα είναι και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερος το κράτος δικαίου, η προσήλωση στο κράτος δικαίου, η προστασία των μειονοτήτων, η παροχή δικαιωμάτων στα, στις μειονότητες κλπ. Γι' αυτό λοιπόν ξεκίνησε η διαδικασία αυτή από το Κοινοβούλιο και οπωσδήποτε θα πρέπει για να έχει κανείς πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια σέβεται πλήρω τι δημοκρατικές αρχές. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Τόμασιτς. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μέλλον αν δεν αναγνωρίσει τα κυρίαρχα δικαιώματα κάθε χώρας να ασκεί αυτόνομη πολιτική σε τομείς που δεν αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης. Ούτε μία υπεύθυνη χώρα δεν ε, θα απειλήσει την ε, εθνική της ασφάλεια μόνο για να ικανοποιήσει τις Βρυξέλλες. Υπάρχουν βέβαια διατάξεις, αλλά μερικοί τις παραπάμπτουν και άλλοι θέλουν να επιβάλλουν ε, τη δική τους ερμηνεία των διατάξεων. Όταν ε, μιλούμε για ανθρώπινα δικαιώματα πολλά και για τα οικονομικά, πολλά, πολλά κρατημέλη παράκαμψαν τους ευρωπαϊκούς κανόνες, ε, αλλά κανένα δεν στυλιτεύθηκε για τον τρόπο ε, που χειρίστηκε τα θέματα αυτά. Ενώ τώρα πολλοί θέλουν να επιβληθούν κυρώσει στην Ουγγαρία και την Πολωνία. Γιατί? Έχει ο κύριος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Όλοι μα, ε, όσοι είναι εδώ εδώ και πολλά χρόνια, παρακολουθούν ε, το πόγκρομ το οποίο έχει εξαπολυθεί εδώ και χρόνια κατά τη ε, Ουγγαρίας. Μπορούμε να πούμε ότι ο κ. Ορμπάν πάντα απαντούσε και εξηγούσε τι δημοκρατικέ του τις πράξεις του με δημοκρατικό τρόπο. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλέ ευθέρετε διαπιστώσει με τι οποίε δεν μπορώ να συμφωνήσω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να λειτουργεί και βλέπουμε ότι τα μέσα ενημέρωση στην Ουγγαρία είναι ακόμα ελεύθερα και πολύ πιο εξελιγμένα και από άλλε χώρε. Υπάρχουν όμω χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που χρησιμοποιούν με διεφθαρμένο τρόπο τους ευρωπαϊκούς πόρους και τολμούν μάλιστα να φυλακίζουν με παράνομο τρόπο τους ε, επικεφαλείς της αντιπολίτευσης. Παρ' όλα αυτά δεν βλέπουμε να γνωρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. ο Επίτροπος Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω σε ορισμένα ζητήματα τα οποία εθίγησαν στη διάρκεια της ε, συζήτησης. Ε, ε, πρέπει να σας πω ότι η Ουγγρική κυβέρνηση αποφάσισε να μην προχωρήσει την διοικητική μεταρρύθμιση. Ωστόσο εγκρίθηκε το Δεκέμβριο η νέα νομοθεσία και προβλέπονται βάσει αυτής τροποποιήσεις εις ε, την δικαστική εξουσία, κυρίως δε εις τον διορισμό των ε, ε, δικαστών ε, και την ε, δυνατότητα ε, να απομακρύνονται χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Αναλύουμε τα νέα νομοθετήματα και λυπούμεθα που λέμε ότι αυτή η μεταρρύθμιση προχώρησε υπερβολικά γρήγορα πριν από την οποιαδήποτε διαβούλευση και πριν την σύμφωνη γνώμη της ομάδας της Επιτροπής της ε, Βενετίας. Ε, είναι ε, γεγονός ότι το δικαστικό, Εθνικό Δικαστικό Συμβούλιο αναλαμβάνει πλέον πολλές εξουσίες και πολλές προκλήσεις. Λόγω αυτών των προκλήσεων έχουν ξεκινήσει διαδικασίες οι οποίες αφορούν, από, έχουν ξεκινήσει από την Επίτροπο κυρία Γιουρόβα, πρωτοβουλίες οι οποίες αφορούν ακριβώς αυτά τα ζητήματα. Ε, Βεβαίω, ακόμα και κάποιες διαθετικές κινήσεις οι οποίες έγιναν ε, στα τέλη τη προηγούμενη χρονιάς ε, δεν ε, αλλάζουν την ουσία των τροποποίησεων που έχουν επέλθει στη δικαστική εξουσία. Την 3η Σεπτεμβρίου του 2019 η απόφαση ενός περιφερειακού δικαστηρίου ε, κρίθη ε, ε, μη σύνομη με το ευρωπαϊκό δίκαιο και στην ε, ε, αιτιολόγηση αναφέρονται ενδεχόμενες ε, πειθαρχικές διαδικασίες καθότι αναφέρεται ότι το, τα εθνικά δικαστήρια θα πρέπει να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στα ευρωπαϊκά, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ε, επίσης ε, υπάρχει ε, το, ο η σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μη διακριτική μεταχείριση και επομένως υπάρχει διαδικασία κατά της Ουγγαρίας και όσον αφορά την διακριτική μεταχείριση ομάδων του πληθυσμού. Θα πρέπει άμεσα η Ουγγαρία να αναλάβει δράση έτσι ώστε να αλλάξει αυτή η κατάσταση να συμμορφωθεί. Θα πρέπει η Ουγγαρία, ε, όπως και όλες οι άλλες χώρες, να έχουν το ίδιο επίπεδο σεβασμού του κράτους δικαίου και των αρχών η Κομισιόν έχει ξεκινήσει και ξεκινάει πάντα ε, εξωτερικούς ελέγχους, audits, οποτεδήποτε ε, προκύπτει ανάγκη για κάτι τέτοιο. Ε, επίσης, η υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίζει ρόλο κλειδί όσον αφορά τις διερευνήσεις τέτοιων κατηγοριών και οπωσδήποτε πρέπει να προστατεύεται ε, ο προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και η χρηστή οικονομική διαχείριση. Ε, ε, στόχος μας πάντοτε είναι η προστασία των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σωστή χρήση τους ε, και οπωσδήποτε η αποφυγή της διαφθοράς. Οι εισαγγελικέ αρχές ελέγχουν την σωστή διαχείριση και την ορθή λειτουργία όλων των διαδικασιών. Θα πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε ε, διαδικασία ή συμπεριφορά η οποία θέτει σε κίνδυνο ε, την χρηστή διαχείριση ε, και των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προκαλεί διασπάθηση ευρωπαϊκού χρήματος. Βεβαίως όλα τα στοιχεία αυτά θα μελετηθούν από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν οι προτάσεις γίνουν δεκτές θα προχωρήσουμε σε ένα επόμενο βήμα. Πρέπει να σας διασφαλίσω, κύριε Πρόεδρε, κύριε βουλευτές, ότι μας ε, ε, ενδιαφέρει και θεωρούμε προτεραιότητα την σωστή λειτουργία του μηχανισμού ε, για την παρακολούθηση του κράτους δικαίου παρακολουθούμε τις ε, εξελίξεις ε, όσον αφορά το κράτος δικαίου, ε, συστηματικές παραβιάσεις ή συστημικά προβλήματα τα οποία μπορεί να μειώσουν την δυνατότητα έκφρασης της γνώμης ή, ή μπορεί να οδηγήσουν σε διασπάθηση η χρήματος και διαφορά, διαφθορά. Τελειώνοντας ε, πρέπει να πω ότι από τη στιγμή που ξεκίνησε η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, παρακολουθούμε στενά τις ε, διαδικασίες και την κατάσταση στην Ουγγαρία. Ευελπιστούμε ότι και με την ευκαιρία της σημερινής συζήτησης ε, η κυβέρνηση της Ουγγαρίας θα μελετήσει προσεκτικά όλα τα θέματα αυτά και θα προσπαθήσει να λύσει οπουδήποτε υπάρχουν προβλήματα. Του Συμβουλίου το λόγο έχει η κυρία Μπρίνιατς. Αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, θα ήθελα και πάλι να σας διαβεβαιώσω ότι η Κροατική Προεδρία και το Συμβούλιο Σύσσωμο αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην τήρηση του κράτους δικαίου και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κοινή μας ευθύνη των κοινοτικών θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών να σεβαστούμε, να προστατεύσουμε και να προωθήσουμε τις κοινέ μας αξίες. Η κρατική προεδρία θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή ε, στις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στη συζήτηση που έγινε. Όπως είπε και ο συγητή, η Φιλανδική Προεδρία τακτικά ενημέρωνε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις διαδικασίες του άρθρου 7 σε σχέση με την Ουγγαρία. Θα ήθελα να επαναλάβω την πρόθεσή μα να συνεχίσουμε αυτή την πρακτική της Φιλανδικής Προεδρίας και η κρατική Προεδρία θα ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις επαφές που θα έχουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις ε, ε, εν λόγω προτάσεις. Ευχαριστώ. Μια πρόταση ψηφίσματος όσον αφορά τις ενεξελίξει ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την Πολωνία και την Ουγγαρία για την περάτωση αυτής της συζήτησης. Η συζήτηση έληξε, η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η δηλώση του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις ανεξελίξει ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την Πολωνία. Εξ ονόματος του Συμβουλίου το λόγο έχει η κυρία Μπρίνιατς. Thank Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, όπως είπαμε προηγουμένως ε, στη συζήτηση για την Ουγγαρία, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα θέματα. Ε, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι αλληλένδετα. Το στρατηγικό μας θεματολόγιο για το 2019-2024 υπενθυμίζει ότι το κράτος δικαίου είναι βασικό εχέγγυο τη σωστή προστασία των κοινών μα αξιών και τη σωστή στήρισή του. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 7, παράγραφο 1 και τη διαδικασία για την Πολωνία που ενεργοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέχρι στιγμή έχουν γίνει τον Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο του 2018 τρει ακροάσει στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Στη συνέχεια, το Συμβούλιο ε, ενημερωνόταν τακτικά για τι εξελίξει στην Πολωνία. Στη διάρκεια του 2019 έγιναν ενημερώσεις ε, για τις εξελίξεις ε, στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων το Φεβρουάριο, Απρίλιο, Ιούλιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο. Η Κροατική Προεδρία θα φροντίσει το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων να συνεχίσει να επιλαμβάνεται το σημαντικό αυτού θέματο. και ταυτόχρονα θεωρούμε ότι η συνεχής διάλογο σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Πολωνίας θα αποφέρει καρπούς. Σήμερα θα κρατήσουμε προσεκτικέ σημειώσει των στοιχείων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και των σχολείων που θα προκύψει στη συζήτηση. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, άξιοι μου βουλευτέ, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο που συμπεριέλαβε στην ατζέντα την κατάσταση σε ό,τι αφορά το κράτο δικαίου στην Πολωνία. Είναι απαραίτητο οι ευρωπαϊκοί θεσμοί να συμβάλλουν στην τήρηση του κράτου δικαίου στο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αντιλαμβάνομαι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθεί στενά την κατάσταση στην Πολωνία και ότι τακτικά ενημερώνεστε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό. Τον προηγούμενο Δεκέμβριο ο Επιτροπό Ρέιντερ είχε την ευκαιρία να ε, ενημερώσει την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Σήμερα η παρέμβαση της Κομισιόν θα επικεντρωθεί στις πιο πρόσφατες εξελίξεις. Να ξεκινήσω με τις εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις 5 Νοεμβρίου του 2019 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με υποστήριξη υποστήριξε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποφάσισε ότι σε ό,τι αφορά το όριο συνταξιοδότησης των ε, τακτικών δικαστών και με την ε, διακριτική ευχαίρεια που τους δίνεται για τη νέα ε, συνταξιοδοτική ηλικία, η Πολωνία έβαλε ουσιαστικά αδικαιολόγητες ε, διακριτικά μέτρα σε ό,τι αφορά τους δικαστές και τη συνέχεια της καριέρας τους βάσει του άρθρου 19.1 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 19 Νοεμβρίου 2019 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εκδόσε επίσης προκρατική απόφαση σε ό,τι αφορά την εξαρτησία του νέου πειθαρχικού σώματος του Ανώτατου Δικαστηρίου. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεώρησε ότι το πολωνικό δικαστήριο θα πρέπει να αξιολογήσει και να αποφανθεί από αυτόν και ότι θα να αποφανθεί κατά πόσον είναι ανεξάρτητο αυτό το πειθαρχικό σώμα της ε, Πολωνίας. Στις 5 Δεκεμβρίου το πολωνικό ανώτατο δικαστήριο βάσει των κριτηρίων που όρισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθη ότι το πειθαρχικό σώμα του Ανώτατου Δικαστηρίου δεν πληρεί τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Δικαίου σε ό,τι αφορά την εξαρτησία των δικαστών και ως εκ τούτου δεν, συμμα... δεν συμμορφώνεται με το κοινωτικό δίκαιο και με το εθνικό δίκαιο. Παρατηρήσαμε μία σειρά αντιδράσεων από τις πολωνικές αρχές που επικρίνουν το, την απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι ο σεβασμός των δικαστικών αποφάσεων με προκαταρτική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι βασική σημασία για την ομοιογενή εφαρμογή του κοινοτικού δίκαιου σε ό,τι αφορά τα πειθαρχικά μέσα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 10 Δεκεμβρίου του 2019, 10 Οκτωβρίου του 2019 αποφάσισε να παραπέμψει το δικαστηρίο σε ό,τι αφορά αυτό το νέο καθεστώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το νέο πειθαρχικό καθεστώς δεν δίνει τις απαραίτητες εγγυήσεις για την προστασία των δικαστών από τον πολιτικό έλεγχο σε ό,τι αφορά τις δικαστικές αποφάσεις. Η κατάσταση συνεχίζεται λοιπόν και εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ σοβαρή. Παρά την προκαταρτική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την απόφαση του Ανατολικού Δικαστηρίου της Πολωνίας, η εφαρμογή των κανόνων αυτών από τους δικαστές ε, υπόκειται κυρώσεις και το πειθαρχικό σώμα εξακολουθεί να λειτουργεί πλήρως. Αυτές οι εξέλιξεις λοιπόν δημιουργούν ένα κίνδυνο μεγάλης ανεπανόρθωτης ζημιάς για τους δικαστές ε, και θα πρέπει τελικά οι τελικές αποφάσεις να λαμβάνονται από ένα ε, πειθαρχικό σώμα το οποίο έχει διαπιστωθεί ότι δεν είναι ανεξάρτητο. Η συνέχιση λοιπόν της λειτουργίας του, του πειθαρχικού σώματος σε, σχέση, σε συνάρτηση και με τις νέες διαδικασίες ε, αυξάνουν την πίεση στο δικαστικό σώμα της Πολωνίας. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κάποιες προτακτικές ε, Αποφάσει και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Για τους λόγους λοιπόν αυτούς, χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει αίτημα εσωτερικών μέσων σε ό,τι αφορά την τρέχουσα διαδικασία επί παραβάση, προκειμένου το δικαστηρίο να αναστείλει την λειτουργία του πειθαρχικού σώματος του Ανώτερου Δικαστηρίου. Τα μέτρα αυτά λοιπόν είναι κατεπήγοντα και θα πρέπει να ληφθούν απαραίτητο στην προκειμένη περίπτωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να συνεχίσει το διάλογο με την Πολωνία σε ό,τι αφορά την κατάσταση για το κράτο δικαίου, σε ό,τι αφορά και την εξέφραση ε, επικοδομητικών λύσεων και την επίλυση του προκειμένου θέματο. Ένα άλλο σημαντικό θέμα, μια πρόσφατη εξέλιξη, έχει να κάνει με ένα νομοσχέδιο σε σχέση με τη λειτουργία του δικαστικού σώματο που συζητιέται από το Πολωνικό Κοινοβούλιο. Το νομοσχέδιο λοιπόν αγγίζει διάφορα στοιχεία όπως η ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος και εξακολουθεί να μα προκαλεί περαιτέρω ανησυχίε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό το, λοιπόν στι 19 Δεκεμβρίου απέστειλα μία επιστολή προ τον Πολωνό Πρόεδρο, στον Πρόεδρο τη Γερουσία και του Κοινοβουλίου, για το νομοσχέδιο αυτό. Ο σκοπό τη επιστολή αυτή ήταν να υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει οι πολωνικέ αρχέ να ενισχύσουν το κράτο δικαίου, προλαμβάνοντα προβλήματα και αντιμετωπίζοντά τα όταν ανακύπτουν. Στην επιστολή, λοιπόν, καλό τις πολωνικές αρχές να διαβουλευτούν με το Συμβούλιο ε, της ε, το Συμβούλιο της Ευρώπη και την Επιτροπή της Βενετίας προκειμένου να μην συνεχίσουν οι διαδικασίε σε ό,τι αφορά το τρέχον νομοσχέδιο, προτού έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Υπογράμμισα στην επιστολή ότι οποιαδήποτε νομοθετική εξέλιξη θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις και την ενόμη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου στην Πολωνία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Γερουσίας ζήτησε γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας που επισκέφθηκε την Πολωνία στις 9 και 10 Ιανουαρίου και θα γνωμοδοτήσει για το νομοσχέδιο. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να ξεκινήσει επικοδομητικό διάλογο σε τακτικές επαφές με τις πολωνικές αρχές με σκοπό να εξευρεθούν ε, επικοδομητικοί τρόποι επίλυσης των ζητημάτων που είναι ανοιχτά. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Προχωρούμε στον κύκλο των ομιλητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Για την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος το λόγο έχει η κυρία Μέτσολα για 1,5 λεπτό. Thank Σας ευχαριστώ. Η θέση της Πολωνίας είναι στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Πολωνία είναι η παλόμενη καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ένταξη της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμανε ότι θα μπορούσαμε να υπερβούμε πέντε δεκαετίες ιστορικού διχασμού και καταπίεσης. Έδωσε ε, ελπίδα στην Πολωνία και ελπίδα στην Ευρώπη. Οι Πολωνοί πολίτες είναι Ευρωπαίοι πολίτες, όπως και οι Πολωνοί δικαστές είναι Ευρωπαίοι δικαστές. Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση γεννά ταυτόχρονα δικαιώματα και υποχρεώσεις και ευθύνες είναι μια δοσοληψία. Υπάρχει δούνε και λαβίν. Έχουμε κοινή ιστορία και θα πρέπει να έχουμε και κοινό μέλλον. Και λόγω αυτού του κοινού μέλλοντος δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηροί όταν ε, το κράτος δικαίου απειλείται στην Πολωνία ή οπουδήποτε αλλού. Δεν μπορούμε να σιωπήσουμε όταν μια εκλογική πλειοψηφία χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για να δικαιολογηθεί το αδικαιολόγητο. Δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηροί όταν η πολωνική δικαιοσύνη τελεί από και δεν πρόκειται να σιωπήσουμε. Ο όρο κράτο δικαίου δεν είναι μια καινή φράση χωρί περιεχόμενο. Σημαίνει ελευθερία, σημαίνει ισότητα, σημαίνει δικαιώματα και σε τελική ανάλυση σημαίνει Ευρώπη. Χωρί την προστασία του κράτου δικαίου, οι συνθήκε μα κινδυνεύουν να μείνουν ωραία λόγια τυπωμένα σε ακριβό χαρτί. Και χωρί μια ουσιαστικά ανεξάρτητη δικαστική εξουσία δεν μπορεί να έχουμε κράτο δικαίου. Και πριν αυτό χαρακτηριστεί ω κομματικό ελιγμό, θα ήθελα να αποσαφηνίσω ότι η υπεράσπιση τη ανεξαρτησία των δικαστών για να ασκούν τη λειτουργία του, χωρί φόβο ή, ή χάρη δεν είναι επίθεση ούτε στο πολωνικό κράτο, ούτε στον πολωνικό λαό. Είναι προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου και σε τελική ανάλυση προστασία του λαού τη Πολωνία. Και θα ήθελα να χαιρετήσω το κουράγιο των πολωνών δικαστών που βρίσκονται εδώ μαζί μα σήμερα. Δεν πρόκειται να σα απογοητεύσουμε, δεν πρόκειται να απογοητεύσουμε την Πολωνία, δεν πρόκειται να απογοητεύσουμε την Ευρώπη. Thank you very much, dear colleague. Our next... Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφε. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία ε, Επίτροπε Γιωρόβα, κύριε Επίτροπε Ρέιντερς, ε, νομίζω ότι είναι σημαντικό ε, να ακούμε τα, εδώ στο Κοινοβούλιο τις καταγγελίες ε, των ε, δικαστών που τους είχαμε εδώ ε, με σάρκα και οστά ε, και ακούσαμε τις καταγγελίες και τα δάκρυά τους. Ε, τα τελευταία δύο χρόνια είδαμε κάποιες προσπάθειες νομοθετικής μεταρρύθμισης που βασίζεται σε αυτήν την καταπατητική κατά κάποιο τρόπο δημοκρατική πλειοψηφία. Δεν είναι δυνατόν κάποια κυβέρνηση που έχει εκλεγεί να θεωρεί τρόπεό της ε, την ε, χώρα ε, από την άλλη πλευρά. Ξέρουμε ότι η Πολωνία ήρθε το 2004 στη μεγάλη διεύρυνση αλλά βασίστηκε, βάσισε το σύνταγμά της στο επαναστατικό σύνταγμα της Γαλλίας και επομένως δεν είναι δυνατόν να επανερχόμεθα συνέχεια και να συζητούμε διαρκώς το δικαστικό σύστημα, τις αποφάσεις ε, των δικαστών, ε, ε, τις αποφάσεις οι οποίες, οι αποφάσεις του Ανατότου Δικαστηρίου της Πολωνίας που αντιτίθενται στα άρθρα 29 και 43 των Ευρωπαϊκών Συνθήκων. Όλα ισχύουν για όλους, συμπεριλαμβανομένης και της Πολωνίας. Ε, ε, είχαμε ε, και την Κυριακή στην Πολωνία μεγάλες διαδηλώσεις των δικαστών, των δικηγόρων με παρουσία και δικηγόρων από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δυνατόν να νομίζουν ότι είναι μόνοι τους. Δεν τους αφήνουμε και δεν μπορούμε να τους εγκαταλείψουμε μόνους τους. Θα πρέπει να έχει κανείς κάποια χώρα δικαίωμα στην χρήση κονδυλίων μονάχα εάν και εφόσον παίζει με τους κανόνες σε του κράτου δικαίου. Ευχαριστώ κύριο Σιμέτσκα. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Όταν ε, οι δικαστές κατεβαίνουν στους δρόμους ε, και διαμαρτύρονται, μπορεί κανείς ε, να υποθέσει ότι πραγματικά συμβαίνει κάτι κακό. Ξέρουμε ότι έχει, έχουν γίνει προσπάθειες εκφοβισμού των δικαστών και ελέγχου των ιδίων. 40 ε, δικαστές, μεταξύ των οποίων κάποιοι βρίσκονται και εδώ, έχουν υπάρξει θύματα οργανωμένων, ενορχιστρωμένων εκστρατιών εκφοβισμού. Ε, η κατάσταση όσον αφορά τους δικαστές ε, δεν έχει ομοιότηση ε, στην ιστορία της χώρας. Δεν είναι δυνατόν να απολύονται δικαστές απλά και μόνο επειδή εφάρμοσαν το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικοστηρίου. Γιατί σε αυτή την περίπτωση τότε τι έννοια έχουν οι κοινέ αξίες και η ευρωπαϊκή δημοκρατία. η Κομισιόν ε, ε, ξεκίνησε με δειλό ενδεχομένω τρόπο, ωστόσο είναι θετικό το ότι ξεκίνησε να ασχολείται με το θέμα. Και όπως είπαμε και προηγουμένως, ε, δεν είναι ένα πολωνικό ζήτημα, γιατί οι Πολωνοί δικαστές είναι Ευρωπαίοι δικαστές και το πολωνικό ζήτημα είναι ευρωπαϊκό ζήτημα και χωρίς ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος δεν μπορεί να υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Η κυρία και έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαι μία εξ αυτών που είχαν την τιμή σήμερα να μιλήσουν με τους εκπροσώπους των ε, Πολωνών εισαγγελέων δικαστών και δικηγόρων και για να σας πω την αλήθεια ακούστηκε μία πρόταση η οποία με εντυπωσίασε ιδιαίτερα στη συνάντηση αυτή θα ήθελα να την επαναλάβω εδώ στο Κοινοβούλιο. Ένας από τους εκπροσώπους είπε ότι